Okay, everybody, if you want to kind of find a seat and settle down and we're going to kick off the first... Καθίστε για να ξεκινήσουμε με το πρώτο πάνελ για τις ε, ημέρες αυτές του 2013. Λέγομαι Μέιτ Μακμάν, είμαι δημοσιογράφος εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά πριν ε, από 20 χρόνια όταν ξεκίνησε αυτό το πρώτο πάνελ ήμουν εδώ, συμμετείχα και το θυμάμαι ακόμα. Και Γνωρίζω δημοσιογράφους λοιπόν από όλη την Ευρώπη και αυτοί όταν βρίσκονται εδώ έρχονται και με βρίσκουν και εγώ πάω και τους βρίσκω. Σήμερα θα μιλήσουμε για νέα κοινωνικά κινήματα, νέα πολιτικά κόμματα και νέες μορφές διαμαρτυρίας στην Ευρώπη με τις εκλογές που θα έχουμε το Μάιο του 2014, 22 με 25 Μαΐου σήμερα για να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση, διότι υποτίθεται ότι θα έχουμε εκπροσώπου από όλε τι πολιτικέ ομάδε, αλλά σιγά σιγά χάνονται. Έχουμε τρει όμω εκπροσώπου. έχουμε την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή εδώ από του Σοσιαλιστέ, την Άννη Ποδηματά, ήταν και η ίδια δημοσιογράφος για αρκετά χρόνια. Εργάστηκε στην ελληνική τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, για Εφημερίδε. Έχει δουλέψει λοιπόν με όλου μα. Σα ευχαριστώ πολύ ε, που είστε εδώ σήμερα. Έχουμε και μια σχετικά νέα ευρωβουλευτή από την Ενωμένη Αριστερά. Ε, είναι η Ίνιας Κριστίνα Ζούμπερ από την Πορτογαλία. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και έχουμε και τον Έντουαρτ Κοσούντσιγκ. Πώς προφέρετε το επίθετό σας, Έντουαρτ. Ο Έντουαρτ λοιπόν είναι ένας πολύ νέος επίσης ευρωβουλευτής έχει κάνει πολύ ωραία βίντεο στο YouTube για να εξηγήσει στον κόσμο πώς εργάζεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, είτε είναι στο τρένο, είτε μιλάει με κόσμο, θα μας πει δυο λόγια αργότερα. Αν δείτε στο Twitter, περιμένουμε ακόμα να έρθει ο κόσμος εδώ στην αίθουσα. Ο λόγος φυσικά για την καθυστέρηση, όπως τα είδατε, είναι οι ουρές που έχουμε για να μπει ο κόσμος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ, πολύ άσχολα τα πράγματα εδώ. Ζητώ συγγνώμη για οποιαδήποτε καθυστέρηση. Πριν δώσουμε το λόγο στους ευρωβουλευτές, ε, ε, μερικές ανακοινώσεις από τον Σεμπάστιαν. Υπάρχουν και άλλε είσοδοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορείτε να μπείτε από το κτίριο Σπινέλη για να μην χρειάζεται να περιμένετε στην ουρά. Όπω σα είπε και ο Έντουαρτ, ε, έχουμε και το Twitter. Μπορείτε να δίνετε, να γράφετε τα tweets σα. Έχουμε και το hashtag CYMD για το σημερινό ε, πάνελ. Λίγο αργότερα θα έρθει και ο Πόν από, το, ε, από την Ευρώπη της Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Θα είναι εδώ σε τρία τέταρτα περίπου. Βρετανός Ευρωβουλευτής. Ήθελα να έρθει σε πέντε λεπτά, αλλά θα είναι εδώ σε 45 λεπτά. Η Τζιν Λάμπερτ από τους Πρασίνους θα έρθει σε δύο, λεπτά, είναι καθοδόν. Και από την Ισπανία, από το ΕΛΚ, ο Αντώνιο Λόπες Ιστουρίς επίσης ε, βρίσκεται σε μία ε, επιμνημόσυνη δέωση για τον πρώην ε, Πρωθυπουργό του Βελγίου, ο οποίος απεβίωσε την περασμένη εβδομάδα. Πρέπει να δώσουμε καταρχάς το λόγο στην Άννη Ποδηματά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα σας καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ε, είπε και η ΜΕΜ, Εγώ και ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπεύθυνη για τα θέματα επικοινωνίας, αλλά και ως ε, δημοσιογράφος ε, για πάνω από 20 χρόνια, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες και έντυπα εν γέννη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σε επαφή με τη νεότερη γενιά. Επιτρέψτε μου να πω με όλο το σεβασμό προς τους ε, άνδρες συναδέλφους, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε πολλές γυναίκες ε, εδώ στην αίθουσα. Όταν ξεκίνησα εγώ πριν από 22 χρόνια, τουλάχιστον στη χώρα μου, και δεν νομίζω ότι ήταν και η μόνη χώρα στην οποία συνέβαινε αυτό, δεν ήταν και προφανές να έχουμε τόσες πολλές γυναίκες στην ενεργό δημοσιογραφία. Ε, χρειάστηκε να δώσουμε μάχη για την πιο ενεργό συμμετοχή των γυναικών, όπως ε, συνέβαινε και εξακολουθεί να συμβαίνει. Ε, με το θέμα της συμμετοχής ε, των, γυναικών στην χάραξη πολιτικής. Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτή τη σύντομη εισαγωγή για το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα να ξεκινήσω από τον τίτλο. Εθνικά προβλήματα, ευρωπαϊκές λύσεις. That we're to deal with. And Είναι ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τόσο ελκυστική. Η Ευρώπη πριν από μερικά χρόνια βρισκόταν σε μια σαφή πορεία προς μεγαλύτερη ολοκλήρωση τότε ήταν αποδεκτό λίγο πολύ από όλους ότι η περισσότερη Ευρώπη ήταν μια πορεία εκ των όνου κάνευ. Η χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική κρίση, συμπεριλαμβανομένων και των απαντήσεων και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση, μας οδήγησε σε εθνικοκεντρικές προσεγγίσεις και ανανεώνησε την διάθεση πολλών να επανέλθουν σε ομιλίες και ρητορικές για την εθνική κυριαρχία, τις οποίες είχαμε ξεχάσει στο παρελθόν και νομίζαμε ότι ήταν στην ιστορία. Τα νέα πολιτικά συστήματα φαίνεται πλέον ότι είναι στη μόδα. Όλο ένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι ελκύονται ε, από εθνικιστικά κινήματα και ομάδες και δεν είναι η αυτή η μορφή των νέων κινημάτων που διαπιστώνουμε και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη μετά την κρίση. Υπάρχουν διάφορες μορφές ε, ατόμων με διαφορετικές ε, απαιτήσεις και δημιουργούν μια νέα Ευρώπη, μια νέα κοινωνία στην Ευρώπη. Υπάρχουν νέα πολιτικά συστήματα των κρατών μελών και της Ευρώπης στο σύνολό τους που είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους. Υπάρχουν οι νέες μορφές συλλογικής έκφρασης, κινήματα, κόμματα, ε, νέες μορφές διαμαρτυρίες. Κάποια από αυτά είναι χαριτωμένα και μάλλον αστεία σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ κάποια άλλα ε, αποτελούν πρόκληση για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα κοινό στοιχείο. Εκφράζουν την απογοήτευση των πολιτών, αν μου επιτρέπετε έκφραση, για το υπάρχον πολιτικό σύστημα και την επιθυμία τους για κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν θα είναι απαραίτητο νέο πολλοί πολίτες ε, είναι ευρωσκεπτικιστές, εκφράζουν τις ενστάσεις τους, τις επιφυλάξεις τους ε, κατά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και τελικώς υπάρχουν και σε βαρές αμφιβολίες ε, και διαμάχες κατά της πολιτικής και των πολιτικών. Οι ενστάσεις, οι επιφυλάξεις νομίζω είναι το βασικό μήνυμα το οποίο μας αποστέλουν όλο ένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες. Έχουμε ένα μήνυμα ε, για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και το θέμα είναι πώς μεταφράζεται αυτό το μήνυμα σε δράση. Εάν συμφωνούμε και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε ότι πολλά από τα σύγχρονα παγκόσμια θέματα, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, των περιβαλλοντικών προβλημάτων, των διεθνών οικονομικών αλλαγών και των κοινωνικών προκλήσεων, χρειάζονται συνολικές και παγκόσμιες λύσεις και επομένως δεν μπορούμε να καθορίσουμε τέτοιες λύσεις σε επίπεδο κρατών μελών εθνών. Συμφωνούμε όλοι νομίζω ότι οι υπερεθνικές ε, δομές και νέες ενώσεις κρατών είναι αυτές οι οποίες θα μας δώσουν αποτελεσματικές λύσεις. Αλλά Μπορούμε να εξετάσουμε αποτελεσματικές λύσεις μόνο σε επίπεδο πολιτών και όχι σε επίπεδο μιας μειονότητας, κάποιων μειονοτήτων, κάποιων ομάδων συμφερόντων ή κάποιων ελίτ. Αυτό λοιπόν είναι τμήμα της μεγάλης ευθύνης που έχουν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η κοινωνία των πολιτών. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να σταματήσουμε τη στήρα απόρριψη και να προσπαθήσουμε να έχουμε δημιουργικά επιχειρήματα και λύσεις. Και αυτό είναι ο ρόλος που τα νέα κινήματα και τα νέα πολιτικά κόμματα πρέπει να διαδραματίσουν κατά την άποψή μου. Για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα η πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη, διότι πρέπει να μάθουν να τίνουν ευήκονους στα όσα έχουν να πούν οι πολίτες. Πρέπει να είναι πιο ανοιχτά, πρέπει να μάθουν, να μάθουμε εμείς, να είμαστε πιο ευέλικτοι πιο διατεθειμένοι να προσαρμοστούμε στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Χρειαζόμαστε ένα νέο συμβόλαιο με πολλές νέες απαιτήσει και να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για τις θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας υπενθυμίζω ήταν και εξακολουθούν να είναι η δημοκρατία, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η ισότητα. Θα πρέπει λοιπόν να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας ε, προς αυτές τις αρχές και αξίες, διότι αυτό είναι περισσότερο απαραίτητο και περισσότερο σημαντικό από ποτέ. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να είναι η σημαντικότερη συνεισφορά των νέων πολιτικών μορφωμάτων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στην ευρωπαϊκή ιστορία. Αυτά λοιπόν εν είδη εισαγωγή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και ε, για όσους δεν ε, το γνωρίζουν, ακόμα και αν μιλήσει αγγλικά, η κυρία Ανυποδηματά είναι αντιπρόεδρος ε, από την, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ελλάδα. Έχετε ερωτήσεις? Έχουμε εκπροσώπους από τις 28 χώρες μέλη της Ένωσης, εκτός από το Λουξεμβούργο. Λοιπόν, να σας θυμίσω πως έχουμε διερμηνία και ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς, αγγλικά, ισπανικά, τσεχικά, πορτογαλικά και ελληνικά, την ε, μετρική γλώσσα της Αντιπροέδρου. Να καλωσορίσω και την Τζιν Λάμπερτ, ευχαριστώ που ήρθες. Ε, εδώ όμως ε, ο Έντουαρντ δείχνει πολύ μοναξιά, μοναχικός. Εγώ θα μιλήσω τσεχικά, γιατί θα είναι πιο απλό για τους τσέχους συναδέλφους. Παρακαλώ βάλτε λοιπόν τα ακουστικά σας και έτσι θα δω και ποιοι είστε Τσέχοι. s čím, s jakým, jako vzkazem mám přijít. Εγώ σκεφτόμουν τι μήνυμα να σας απευθύνω σε αυτή τη συνεδρίαση. Σκεφτόμουν, σκέφτηκα λοιπόν τη ζωή μου και ίσως θα είναι καλό να, να χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα. Σήμερα είμαι 42 χρονών. Και Έχω ζήσει πολύ μεγάλες αλλαγές από την άλλη πλευρά του σιδηρού παραπετάσματος. Όταν ήμουν 19 ετών έφυγα από την κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία τότε και ζήσα, όπως καταλαβαίνετε, για 19 χρόνια σε ένα καθεστώς που, που δεν υπήρχε ελευθερία. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι της ζωής μου. Στο δεύτερο κομμάτι της ζωής μου μπόρεσα να ταξιδέψω σε ολόκληρο τον κόσμο και να γνωρίσω νέους από διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς και γλώσσες. Έβαλα σήμερα ένα ωραιότατο μαύρο μπλουζάκι που αγόρασα πριν από πολλά χρόνια στα νησιά Καλάπαγκος, πριν να γίνω ευρωβουλευτής και ίσως από πρώτης ματιάς ε, να μοιάζει με το Τζέκι Βάρα η φωτογραφία που έχω πάνω στο μπλουζάκι μου, αλλά δεν είναι. Είναι μια εικόνα του Καρόλου Δαρβίνου, γιατί το μπλουζάκι το πήρα στα Γκαλάπαγκος και τώρα δεν θα πω ποιος από τους δύο συνέβαλε περισσότερο στην ιστορία του ανθρωπίνου είδους αλλά να πω για την εξέλιξη, την επανάσταση και την ταχύτητα να προσθέσω εγώ. Εάν δούμε, εάν δει κανείς την ιστορία του ανθρωπίνου είδους, πάντοτε βλέπουμε διάφορες φάσεις, βλέπουμε την εξέλιξη των όντων, πιστεύουμε και ότι οι αλλαγές αυτές ε, οδεύουν προς το καλύτερο, αλλαγές οι οποίες ε, σταδιακά γίνονται, περνούν γενναίες μέχρι να εμπεδοθούν και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι όταν ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα, όταν ας πούμε παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κατάφορα, οδηγείται ο κόσμος σε επανάσταση. Εγώ έζησα την πολιταρχική κοινωνία και έζησα και την επανάσταση. η οποία ακολουθεί μάλλον φυσιολογικά. Η ζωή δεν είναι άσπρο μαύρο, η ζωή είναι πολύχρωμη. Και νομίζω πως όλοι μπορούμε να δούμε πως η Ευρώπη έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία 15 χρόνια και θα συνεχίσει να αλλάζει. Βλέπετε και στο Twitter τα μηνύματα που μας στάνουν εδώ στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να βρείτε έναν χάρτη που δείχνει πώς άλλαξε η Αθήνα τα τελευταία χίλια χρόνια. Προσπαθήσω να το προβάλλω τώρα, θα το δείτε σε ένα λεπτάκι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι 50 χρόνια εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ιστορίας, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποιες ε, ομάδες του πληθυσμού που προτιμούν τις επαναστάσεις, ενώ υπάρχουν κάποιες άλλες ομάδες ε, του πληθυσμού, του ευρωπαϊκού, που προτιμούν την ε, φυσιολογική εξέλιξη στην πολιτική, όμως είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άρα πρέπει να μιλήσουμε για πολιτική. Στην πολιτική έχουμε να κάνουμε με επιχειρήματα, να δούμε που υπάρχει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε διάφορες ομάδες ανθρώπων. Να διακρίνουμε τις επιθυμίες του κόσμου. Αυτό το οποίο έχει χαθεί στην πολιτική ίσως είναι αυτός ο αγώνας για ελευθερία και τα μεγάλα ε, καθιερωμένα παραδοσιακά κόμματα ε, γίνονται πιο συγκεχημένα και αναπτύσσονται περισσότερα εναλλακτικά κόμματα δεξιά και αριστερά δυστυχώς κάποιες φορές με πολύ ακραίες απόψεις. Το πρόβλημα στην Ευρώπη και στην τσεχική δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ότι η διαχωριστική γραμμή δεν είναι ελευθερία και μη ελευθερία, αλλά κοινωνικά συμφέροντα ορισμένων κοινωνικών ομάδων. Διατήρηση δηλαδή του status quo, αυτού που οι περισσότεροι θέλουν να υποστηρίξουν ως κοινωνικό του status. Και πάλι, και βλέπω και άλλα μηνύματα Twitter και να αναφερθώ σε αυτό το χάρτη που έβαλα πριν από, σας έδειξα πριν από λίγο, να σας δείξω δηλαδή πώς έχει αλλάξει η Ευρώπη τα τελευταία χίλια χρόνια. Σας ευχαριστώ. <clears throat> Ehm, ah, και τώρα να δώσω το λόγο στην Τζιν Λάμπερτ. Έχεις ε, με ένα γαλλικό όνομα, αλλά είσαι από το Essex και είσαι μέλος του Πράσινου κόμματο, τη Αγγλία και τη Ουαλίας. Είσαι από το 99 εδώ ω και αντιπρόεδρος σήμερα των ε, Πρασίνων και ήδη από τη δεκαετία του 70 είχε μπει στο κόμμα το οικολογικό και εδώ ασχολείσαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Επιτροπή Απασχόληση, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είσαι και ακτιβίστρια, ιδιαίτερα ενεργή. Με <laughs> όλα αυτά που είπες μου θύμισες πόσο καιρό είμαι εδώ. Βλέποντας το, το, το, θέμα για αυτήν εδώ τη συζήτηση, να πω ότι κάτι που θέλω να πω εξ αρχής είναι ότι αυτή η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως λύση των προβλημάτων δεν είναι κάτι το νέο και εξαρτάται πολύ από το πού βρίσκεται κανείς, από πού κοιτάει την εικόνα. Από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τη δικό μου πολιτικό, πολιτική ιστορία υπήρξε φάση όπου όντω θεωρούσαμε πως θα ήταν η λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση ω το σώμα το οποίο εξέταζε την περιβαλλοντική ε, πολιτική πολύ σοβαρά και προσέφερε περισσότερο όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα δικαιώματα στην εργασία, ενώ σταδιακά έχει υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση για, ε, για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ήταν πρόβλημα βέβαια για όσους θεωρούσαν ότι η αγορά ήταν ο βασικός παράγοντας, ότι ήταν αυτό το οποίο θα συνένωνε την Ευρώπη και θα βοηθούσε να διατηρηθεί αυτός ο ρυθμό, η ειρήνη ως βάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όσοι λοιπόν το είδαν ε, ότι ήταν ε, η βάση για την αγορά, για την ελευθερία, την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, ήρθαν σε κάποια ένταση με αυτούς που έχουν τόσο, τόσο αυτή διαφορετική πολιτική άποψη. Αυτή τη στιγμή βέβαια το θέμα είναι η ελεύθερη κυκλοφορία, η τέταρτη ελευθερία που θεωρώ πως πάντοτε είναι η πιο, αυτή που αμφισβητείται περισσότερο ε, ε, για τον κόσμο που ζει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ ο κόσμος ε, το θεωρεί την πιο πολύτιμη ελευθερία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα ήταν δύσκολο να, να ισχυριστεί κανείς για όσους βλέπουν ως μια προοδευτική δύναμη. Όταν αν δει κανείς πώς χειριστήκαμε την κρίση, αυτό ε, υπονομεύει την άποψη όσων θεωρούν πως η Ευρώπη έχει ένα όραμα και μάλιστα ένα θετικό όραμα για το μέλλον. Έχουμε προβλήματα όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης βέβαια και Γίνεται όλο ένα και περισσότερος αγώνας για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι δεν είναι μόνο οικονομική η κρίση, είναι και κλιματική η κρίση. Και σε αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να ενεργεί η Ευρώπη και πολύ πιο δραστήρια. Τι γίνεται λοιπόν με όλα αυτά τα κοινωνικά κινήματα τα οποία αναπτύσσονται και ποιος είναι ο αντίκτυπος. Όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχουν κάποιε πολύ, μορφές, πολύ παλιές μορφές πολιτικής και πολιτικών κινημάτων. Θα έλεγε κανείς ότι σε αυτή τη στιγμή έχεραν μιας ε, χρυσής εποχής ότι υποστηρίζουν τις θεμελιώδεις αξίες ε, και ο κόσμος ε, είχε ίσως κάποια εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα, ενώ βλέπουν αυτή τη στιγμή ε, ότι αυτή είναι το πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη στο να αναπτύξουν ιδέες που να ωφελούν τον κόσμο γενικότερα. Αυτή η κομματική πολιτική θεωρείται λοιπόν πλέον λιγότερο ικανή, λιγότερο ευέλικτη, προσαρμόσιμη και βέβαια οι ίδιοι θέλουν να διατηρήσουν το status quo, ενώ στην ουσία θέλουν να διατηρήσουν κάποιο είδους σταθερότητα, ώστε να μην υπάρξει μια, ένα εφέ ντόμινο προς κάτι άλλο άγνωστο. Το ότι ο κόσμος βλέπει ότι όλοι οι πολιτικοί κοιτάνε τον εαυτούλη τους, αυτό δεν είναι συμπέρασμα ή απόφθηγμα λόγω της κρίσης. Υπήρχε ανέκαθεν αυτή η τάση και βλέπουμε όλο, όλο ένα και περισσότερους νέους να μην θέλουν ή να μην σκέφτονται να πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν θέλουν να ασχοληθούν ούτως ή άλλως με την πολιτική. Και νομίζω πως κάνουμε λάθος αν πιστεύουμε πως αυτό είναι ένα μήνυμα πολιτικής απάθειας. Είναι ένα μήνυμα μάλλον ότι πολλοί θέλουν να κάνουν κάτι το τελείως διαφορετικό. Θέλουν δηλαδή να κάνουν πολιτική ανάλογα με θέματα και όχι κομματικά. Και αυτό έχει τα πλεονεκτήματά του, αλλά έχει και τα μειονεκτήματά του. Γιατί όλοι όσοι έχουμε συμμετάσχει σε πολιτικά κινήματα, σε κάποιο στάδιο της ζωής μας γνωρίζουμε πως είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς πολιτική για ένα μόνο θέμα. Δηλαδή όταν ζητά μόνο ένα πράγμα. Αλλά ότι είναι και πάρα πολύ εύκολο να κάνεις και πολιτική αντιπολίτευση. Όταν ξέρεις δηλαδή τι δεν θέλεις. Ενώ είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις πολιτική όταν πρέπει να συνδέσεις όλα αυτά τα κομμάτια και να δεις ακριβώ τι θέλεις να κάνεις και τι θέλεις να υποστηρίξεις και τι αλλαγές θέλεις να γίνουν στον κόσμο. Τα κοινωνικά κινήματα λοιπόν που συντεριάζουν μέσα σε αυτή τη φάση κρίσης, να αναφέρω ένα-δύο παραδείγματα. Το ένα θα είναι, είναι το Occupy. Το κίνημα Occupy και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό χώρο ώστε να μπορεί κανείς να μιλήσει για την οικονομία και τι θέλει να κάνει η οικονομία πώς θα πρέπει να δικούνται οι τράπεζες και ποιος είναι ο στόχος της οικονομίας. Γίνεται λοιπόν ένας προβληματισμός για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Είναι μια διαδικασία που είχε πραγματικά αντίκτυπο, πιστεύω, γιατί υπάρχει κόσμος που πραγματικά θέλει να μιλήσει για την ουσία, για τη βάση, για τα θεμέλια με βαθύ τρόπο και αυτό ε, είχε σχέση και με τα όσα συμβαίνουν ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου δηλαδή υπάρχει αυτή η δημόσια δυναμική ε, και η οποία έχει οθήσει και την πολιτική δυναμική εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ακόμα αγωνιζόμαστε προσπαθούμε να ε, βρούμε αυτή τη σχέση και αυτή τη σύνδεση, η οποία ωστόσο είναι ισχυρή και συνεχιζόμενη. Ένας από τους άλλους τομείς που ίσως θα πρέπει να αναφέρω εν συντομία είναι η εκστρατεία online και να μιλήσω για το Άβας Πρόκειται για, εκείνη, για εκείνο το κίνημα για την εμπορική συμφωνία για τα εμπορικά σήματα. Από τη μια πλευρά έχουμε ένα πολύ και μια πολύ βαρετή και τεχνική συμφωνία η οποία όμως έχει τεράστιο αντίκτυπο και κανονικά ο κόσμος δεν ασχολείται όμως με όλα αυτά. Είναι πολύ δύσκολο, άστο για τους ειδικού, λέει συνήθως. Αλλά το γεγονός ότι έγινε ε, online εκστρατεία με κόσμο ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αφοσιωμένος και γνώστης των θεμάτων και βρήκε και τρόπο για να έρθει σε επαφή με το ευρύ κοινό ε, όσον αφορά την ε, κοινοποίηση των θεμάτων και την ποινικοποίηση ορισμένων υποθέσεων Έφτασε στο Κοινοβούλιο το θέμα, ε, τέθηκαν θέματα για τη διαφάνεια, για το περιεχόμενο, για τις επιπτώσεις όλων αυτών και έτσι μετετράπησε ένα πολιτικό ζήτημα το όλο θέμα με το οποίο έπρεπε να ασχοληθούν οι βουλευτές και τελικά ε, απορρίφθηκε το, η συμφωνία αυτή. Ορισμένοι από εμά θεωρούμε πως ήταν το σωστό αυτό, το επιθυμητό. Πιστεύω πάντως ότι η πραγματική συμμετοχή του κόσμου είναι αυτή που σημαίνει τη διαφορά. Να είναι κανείς δηλαδή πρόθυμος να συμμετέχει και να ασχολείται με τα θέματα. Αυτό δείχνει μια μετακίνηση. Τώρα τι θα σημαίνει για τις εκλογές θα δούμε. Μπορεί ε, ο κόσμος να θεωρήσει πως έκανε αυτό που έπρεπε από πολιτικές άποψεις ε, για το θέμα και τα τα λοιπά μπορεί να μην θεωρήσουν ότι πρέπει να βγουν από το σπιτάκι τους στις 22 Μαΐου και να πάνε να ψηφίσουν. Πάντως είναι ένας τρόπος για πραγματική πολιτική δέσμευση που έχει αντίκτυπο. Αυτά ήταν ένα-δύο παραδείγματα, υπάρχουν και άλλα βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις και για σας, όπως και τους <laughs> πολύπους ε, στο πάνελ. Εσύ ασχολείσαι με, τα, με το Twitter. Έχεις κάποια ενδιαφέροντα tweet που θα ήθελες να μας ε, διαβάσεις αυτή τη στιγμή. Είχαμε για παράδειγμα την ανάδυση αυτών των νέων ε, ακραίων ομάδων, αν η πολιτική πλέον δεν έχει τόσο μεγάλη σχέση για την Ευρώπη. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε κατά νου τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που δίνονται. Να δώσω τώρα το λόγο στην Πορτογαλίδα Ευρωβουλευτή, την ε, Ινιές Κριστίνα Ζούμπερ. Είναι αντιπρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων. Ήσασταν μέλος του Πορτογαλικού Κομμουνιστικού Κινήματος, έτσι. Θα μιλήσετε πορτογαλικά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα μιλήσω πορτογαλικά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για τη διοργάνωση και για την πρόσκληση. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πολύ και είναι το θέμα της διαμαρτυρίας. Εγώ εκλέγομαι με το Πορτογαλικό Κομμουνιστικό Κόμμα που υπάρχει ε, εδώ και 100 χρόνια. Είμαστε δύο εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, εγώ που είμαι 33 ετών και άλλο ένα μέλος το οποίο έχει, ε, είναι 34 χρονών. Το κόμμα μας υπάρχει από το 1921 και ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο αντιστάθηκε διαρκώς ε, κατά τη διάρκεια των χρόνων του φασισμού στην Πορτογαλία και που συνέβαλε στο να υπάρξει η δημοκρατική επανάσταση στη χώρα μας. Και γι' αυτό το λόγο το θέμα της αντίστασης και της διαμαρτυρίας είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα παρόν ε, στις ζωές μας. Ήθελα να σας πω πως ε, τη σήμερα ημέρα το θέμα της ε, διαμαρτυρίας στη χώρα μου, την Πορτογαλία, έχει άμεση σχέση με τη διαμαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να είναι αλλιώς, διότι άλλο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στα λόγια και άλλο είναι το τι, πώς επηρεάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη ζωή των, άμεσα των ανθρώπων και για τη χώρα μου η Ευρώπη είναι μια τρόικα η οποία έχει επηρεάσει πολύ συγκεκριμένα την καθημερινή ζωή του κόσμου. Και με αυτή την έννοια δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίσει κανείς αυτές τις διαμαρτυρίες από τις διαμαρτυρίες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό γιατί για μένα, για παράδειγμα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το να βλέπω το τι γίνεται εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για την κοινωνική Ευρώπη, το κοινωνικό πρότυπο και την κοινωνική εξέλιξη και εκείνο που οι τεχνικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν στη χώρα μου. Αυτό που έκαναν στη χώρα μου πριν από τρία χρόνια ήταν να επιβάλλουν φυσικά με την ε, συνενοχή των κυβερνήσεων την ε, ε, φτώχεια για τον κόσμο. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή παραδόξως οι άνθρωποι ε, αρπάζονται από τα εθνικά του συντάγματα για να υπερασπιστούν τα κοινωνικά τους δικαιώματα που είναι και εκτιμένα και τα εργατικά τους δικαιώματα που είναι και εκτιμένα και ότι κατά κάποιο τρόπο έτσι προσπαθούν να αμυνθούν κατά των επιθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω, να δώσω, να κρίνω οτιδήποτε έτσι, απλώς ε, κάνω διαπιστώσεις για να καταλάβουμε αυτήν την ε, διχοτομία που υπάρχει ανάμεσα στο τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τι είναι για τον απλό κόσμο. Αυτές οι διαπραγματεύσεις, ας πούμε, οδήγησαν στο να καταργηθούν τα επιδόματα Χριστούγεννων διακοπών, τη μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση διαφόρων εργατικών δικαιωμάτων ώστε να διευκολυνθούν οι απολύσει, την ε, επέκταση του ωραρίου εργασίας, την καταστροφή πολλών ε, δημοσίων υπηρεσιών όπως τα νοσοκομεία, όπως ε, τα κέντρα υγείας, ιδιωτικοποίησαν βασικές δημόσιες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα τα ταχυδρομεία και που τώρα μειώνονται μέσω αυτών των ιδιωτικοποιήσεων, οι οποίες συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα λοιπόν δεν έχει νόημα να λέμε ναι, ναι, αλλά θα έρθουν χρήματα για την Πορτογαλία ε, τα επόμενα χρόνια, γιατί γνωρίζουμε ότι μόνο τους τόκους των δανείων να μπορέσουμε να πληρώσουμε είναι περισσότερα τα χρήματα από τα χρήματα που θα πάρουμε τα επόμενα 7 χρόνια. Μα είναι φυσιολογικό να, έχουν επαναστατήσει, να έχει επαναστατήσει ο κόσμος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πιστεύω και πρόκειται για δική μου ανάλυση, πιστεύω πως το κίνημα διαμαρτυρίας της Πορτογαλίας έχει συγκεκριμένα πορτογαλικά χαρακτηριστικά και είναι ένα κίνημα το οποίο είναι τακτικό, είναι ειρηνικό και αυτό έχει να κάνει και με την ε, διαδικασία της Επανάστασης του 1974. Έχουμε συνδικαλιστικό κίνημα πολύ ισχυρό, αλλά ε, θα πρέπει να δούμε ότι τι γίνεται με, όχι μόνο στις μεγάλες διαδηλώσεις που γίνουν στη Λισαβόνα ή στο Πόρτο ε, με πολλές χιλιάδες κόσμο, αλλά και για όσους οργανώνονται και γύρω και από ε, συγκεκριμένο οργάνωση, για το κέντρο υγείας που θα κλείσει στην τάδε περιφέρεια ή για τις θέσεις, ε, ε, ή μάλλον για τα χειδρομεία που θα κλείσουν σε, κάποιο απομακρυσμένο, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, αντιδρά ο κόσμος. Πρόκειται για κινήματα, ας πούμε, του κόσμου κατά της αύξησης του κόστου των ε, δημόσιων μεταφορών. Δεν είναι, δηλαδή δεν βλέπει κανείς την διαμαρτυρία μόνο στις μεγάλες διαδηλώσεις αλλά και γύρω από μικρές ε, και τοπικές διεκδικήσεις. Ήδη γίνανε δύο μεγάλες ε, γενικές απεργίες στην Πορτογαλία με μεγάλη επιτυχία. Κάναμε, ήταν διαδηλώσεις που δεν είχαμε δει ποτέ και είναι ένα φαινόμενο ενδιαφέρον. Είμαστε ναι, μεν ένα συνδικάτο οργανωμένο και έρχονται, έρχεται κόσμος ο οποίος ποτέ δεν είχε συμμετέχει σε διαδήλωση στη ζωή του, ποτέ δεν είχε οργανωθεί σε συνδηλικανιστικό κίνημα ούτε σε κοινωνικό κίνημα, αλλά που αυθόρμητα τώρα ε, προσέρχεται για αυτές τις διαμαρτυρίες. Και επίσης υπάρχει κάτι το οποίο θεωρώ πως είναι πολύτιμο για τους δημοσιογράφους και αναλύονται σήμερα εκείνα τα κινήματα τα οποία κινητοποιούνται μέσω του ίντερνετ, του facebook και του twitter κτλ. Είναι αλήθεια πως αυτά τα κινήματα είχαν πολύ μεγάλο αντίκτυπο, δηλαδή ε, κινήματα που ξεκινάνε από ε, μια ομάδα στο facebook ας πούμε και αυτό πολύ συχνά συμβαίνει γιατί ο κόσμος δεν θέλει να συνδέεται με κάποιο πολιτικό κόμμα και αυτό είναι αλήθεια ότι η αποτροπή προς την πολιτική ε, ε, ε, προκύπτει από αυτήν την σύγχυση, από αυτήν την απογοήτευση απέναντι στις πολιτικές υποσχέσεις που έγιναν αλλά που δεν τηρήθηκαν. Πιστεύω πως ο κόσμος δεν πιστεύει πια στην πολιτική και αυτοί που φταίνε είναι οι κυβερνήσεις. Αυτοί φταίνε, οι κυβερνήσεις φταίνε για την απογοήτευση του κόσμου. για να τελειώσω αυτό που έλεγα για τα κινήματα μέσω του ίντερνετ. Είναι παράξενο γιατί αυτοί, αυτά που ξεκινάνε από το ίντερνετ ε, αγνοούν τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή τον τύπο που ε, ως αρχή μετά αυτά τα μέσα παίρνουν και δημοσιοποιούν περισσότερο ε, τι, το τι συμβαίνει και πολλαπλασιάζουν τον αντίκτυπο. Για παράδειγμα, εγώ δεν έχω Facebook. και ενημερώθηκα για αυτές τις διαδηλώσεις μέσω της τηλεόρασης. Δηλαδή ξεκινά η, η σπίθα από το ίντερνετ, αλλά μετά η φωτιά εξαπλώνεται από τα, από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης που παίζουν καθοριστικό ρόλο και σε αυτή την περίπτωση. Να σας πω δε ότι αυτό το Σάββατο θα γίνει μια διαδήλωση και, για να περάσουμε την γέφυρα της 25ης Απριλίου που είναι μια γέφυρα στην, της Λισαβόνας. Το Υπουργείο απαγόρευσε αυτή τη διαδήλωση. Πρώτη φορά, έχουμε δημοκρατία, είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση απαγορεύει διαδήλωση. Για το δικαίωμα σε συγκέντρωση και σε διαδήλωση είναι ε, ε, ιερό και όσιο. Ε, επικαλέσει και θέματα ασφάλειας. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο διαμαρτυρίας όπου η κυβέρνηση προσπαθεί να ποινικοποιήσει και να απαγορεύσει τις διαμαρτυρίες μας. Ε, αυτή η διαμαρτυρία θα γίνει λοιπόν την το, το, το Σάββατο Τι θα κάνει ο κόσμος λοιπόν, θα περάσει με τα λεωφορεία γιατί τους απαγορεύθηκε να περάσουν περπατώντας. Θέλαμε να υπάρξει αντίκτυπος και στις αστυνομικές δυνάμεις και στους ε, διαδηλωτές. Θέλουμε λοιπόν ο κόσμος να καταλάβει τους λόγους για τους οποίους ε, αγωνιζόμαστε. Κάτι ακόμα να πω όσον αφορά την άκρα δεξιά. Στην Πορτογαλία ευτυχώς δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο, όπως στην Ελλάδα για παράδειγμα. Δεν το έχουμε γιατί η ιστορία μας είναι διαφορετική. Εγώ όμως ε, ήθελα να πω κάτι που νομίζω ισχύει για όλους το φαινόμενο των ε, εξτρεμιστικών ομάδων, γιατί ακριβώς υπάρχουν καταρχήν. Γιατί τους αφέθηκε χώρος για να, ε, για να υπάρξουν. Γιατί ο κόσμος σήμερα είναι σε μια κατάσταση όπου είναι απαραίτητο αυτή, αυτό το είδος των ομάδων που κάνουν από ε, ε, τράγους τους μετανάστες και τα λοιπά. Δημιουργήθηκε χώρος για να δημιουργηθούν γιατί οι κυβερνήσεις ήταν ανίκανες να καλύψουν τα προβλήματα, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να δώσουν την αξιοπρέπεια που χρειάζεται να έχουν αυτές, να έρχει ο κόσμος και γι' αυτό και αυτές οι ομάδες έχουν ε, συμπάθεια ακόμα και από ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα, καμία σχέση με τα ακροδεξιά κινήματα. Να, είναι πολύ σημαντικό ωστόσο να μην αφήσουμε με την ε, δικαιολογία ότι οι ακροδεξιές ομάδες αυτές που εμφανίζονται στην Ελλάδα αλλά και αλλού, στη Γαλλία ας πούμε, πρέπει να τους καταπολεμήσουμε, αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην γίνει κανένας είδους ε, ε, σύγχυση με τις διαμαρτυρίες που κάνει ο κόσμος για να υπερασπίσει τα δικαιώματά του. Να μην ε, δηλαδή θεωρηθεί αποδειχθεί ότι αυτές οι διαμαρτυρίες είναι εγκληματικές ενέργειες όπως αυτές των ε, ακροδεξιών κομμάτων. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μόλις ήρθε και ο Ισπανός Ευρωβουλευτής πάνω στην ώρα. Μόλις ήρθε και ο Αντώνιο Λόπεθ ε, Ιστουρίς ε, White, είναι από το ΕΛΚ, τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην Ισπανία φυσικά είναι στο Παρτίδο Ποπουλάρ Εδώ συμμετέχει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και είναι και αναπληρωτής ε, στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Ασχολήθηκε με την πολιτική αποφοιτητής την ε, ε, Ένωση των ε, Νέων Γενεών, Νουέβας γενερασιών, που ήταν το κίνημα νέων του Παρτίδο Ποπουλάρ στην Ισπανία, συνεργάτης του Αθνάρ. Σα ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σα παρουσία εδώ και σα δίνουμε αμέσω το λόγο. Εν τω μεταξύ μπορείτε να προετοιμάσετε τι ερωτήσει σα, διότι το σκεπτικό μα είναι να κάνουμε συζήτηση φυσικά. για λόγους ε, διερμηνίας ε, θα μιλήσω ισπανικά. Ε, φορέστε τα ακουστικά σας λοιπόν. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη από τους διοργανωτές και από όλους εσάς για την καθυστέρησή μου. Όπως θα γνωρίζετε, την περασμένη ομάδα απεβίωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Βίλφριντ Μάρτενς, και αυτή την εβδομάδα ε, έχουμε διάφορες ε, τελετές ε, για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτού του τόσο σημαντικού Ευρωπαίου και πέραν της κηδείας η οποία θα γίνει το Σάββατο εδώ στις Βρυξέλλες έχουμε και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. ήθελα να αναφέρω τον Βίλφρεντ Μάρτες, διότι και για εμάς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και για όλους όσους ασχολήθηκαν με το ευρωπαϊκό όραμα, ήταν παράδειγμα για τη μάχη κατά της αδιαφορίας, κατά της έλλειψης πληροφόρησης ε, που έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να τιμήσω τη μνήμη αυτού του ανθρώπου, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια έδωσε μάχη, ώστε να είμαστε όλοι εμείς εδώ να μιλούμε και να συζητούμε για την Ευρώπη, για τα ελαττώματά της, για τα, υπερτε... Ε, για τα ε, καλά τη στοιχεία και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για το θέμα αυτό στο μέλλον ε, μέσα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Για να είμαι σύντομος, διότι ξέρω ότι θα έχουν ε, σίγουρα πει αρκετά πράγματα οι συνάδελφοι και για να δώσω χρόνο για περισσότερες ερωτήσεις και συζήτηση, να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βλέπει τις επόμενες ευρωεκλογέ με λίγο διαφορετικό πνεύμα. Η συνθήκη, όπως γνωρίζετε, δίνει στις ε, πολιτικές ομάδες και στα πολιτικά κόμματα και χαίρομαι που όλοι πλέον συνεργαζόμαστε και μπορούμε να παρουσιάσουμε κοινέ ιδέες για τον υποψήφιο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε ότι πλέον οι συνθήκες ε, δίνουν τη δυνατότητα να ε, ψηφίζεται ο πρόεδρος από, την, από τους πολίτες. Πρέπει να γίνει λοιπόν μια ευρωπαϊκή πολιτική συζήτηση πέραν της συζήτησης που γίνεται σε εθνικό επίπεδο, διότι ένα από τα προβλήματα που υπάρχει ακριβώς λόγω της έλλειψης ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το γεγονός ότι δεν συζητούνται επαρκώς οι ευρωεκλογέ. Εσείς και εσείς ως δημοσιογράφοι το γνωρίζετε, πάντα το 90% της συζήτησης για τις ευρωεκλογέ επικεντρώνεται σε εθνικά θέματα και έτσι οι πολίτες δεν είχαν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις ευρωεκλογέ. Αυτή λοιπόν η ασήμαντη υπόθεση των ευρωεκλογών ε, μεν, αλλά την τόσο σημαντική στην πραγματικότητα μέσω και τις εκλογές του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι μια μοναδική ευκαιρία ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε όλοι ανοιχτά με διαφάνεια, ώστε να γνωρίσουν όλοι οι πολίτες τι ακριβώς είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τι μπορεί να τους προσφέρει. Εάν πρέπει να κάνουμε και αυτοκριτική ή επικρίσεις στη διάρκεια αυτής της συζήτησης ή να ακούσουμε τους πολίτες για να μας πούνε τι θέλουν, αυτή η συζήτηση είναι αυτή η οποία θα πρέπει να γίνει το 2014 από όλους μας, ακόμα και για αυτούς που έχουν αμφιβολίες για το οικοδόμημα και για όλους όμως ε, όσους πιστεύουν ακράδαντα σε αυτό. Κατά την άποψή μου θα πρέπει όλοι να τηρήσουμε μια επικοδομητική στάση. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα ε, γιατί ε, θέλουν να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εγώ θεωρώ ότι πάντα πρέπει να ακούμε και αυτούς οι οποίοι έχουν αμφιβολίες και να πρέπει να τους δίνουμε παρκή στοιχεία, διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχουν όλοι αρκετή ενημέρωση. Και έτσι τι έγινε. Θεωρείται δευτερεύον ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κράτη-μέλη, ε, νομίζω επειδή υπάρχει και μία ε, διαμάχη μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και κρατών μελών, που κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να υπάρχει, οδήγησε λοιπόν σε ε, εκλογές ε, οι οποίες για παράδειγμα, όταν γίνονται σε μια μεγάλη χώρα, θεωρούνται ότι παραλύουν την δυνατότητα λήψη απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει την πορεία. Εμεί όλοι είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν συνέβαινε αυτό σε προηγούμενε θητείε, σε προηγούμενε προεκλογικέ εκστρατείε και χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει δράση σε θέματα επικοινωνία. Ε, καλεί όσο το δυνατόν περισσότερο δημοσιογράφο, διότι όλοι εσεί είστε δημοσιογράφοι και είστε το μέσο επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαίους πολίτες. Και νομίζω και φαντάζομαι και πιστεύω ότι οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι χρήσιμο, ανταγωνιστικό και θα πρέπει να είναι παρούσα στο ε, παγκόσμιο περιβάλλον. Πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτές τις πολιτικές που είχαμε σε εθνικό επίπεδο στο παρελθόν, πλήρους απουσίας των ευρωπαϊκών θεμάτων. Ε, δεν ξέρω, πολλοί συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο στην πολιτική, είτε από το κόμμα μου, είτε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το ή οτιδήποτε, τίνουν όταν κάτι είναι καλό να λένε ότι είναι δική τους πολιτική και όταν είναι κάτι κακό να ρίχνουν το φταίξιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, χρησιμοποιούν πολύ συχνά οι πολιτικοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και στη χώρα μου και σε πολλές άλλες ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλες μάλλον. Εμείς νομίζω ότι δημιουργούμε κάτι το οποίο είναι αξιοζήλευτο εκτός των συνόρων μας. Εγώ λόγω των καθηκόντων μου έχω επαφές με τη Λατινική Αμερική, με την Αφρική, με την Ασία και ανέκαθεν εξέταζαν με μεγάλο, έβλεπαν με μεγάλο ζήλο το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί από την Αλγερία, από το Μαρόκο, από την Τινησία μου έλεγαν ότι αν είχαν αυτή το 1 δέκατο αυτών που έχουμε καταφέρει εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να λύσουν πάμπολα προβλήματα στην περιοχή τους. Τώρα που η Αραβική Άνοιξη ε, διανύει τόσο δύσκολη περίοδο. Ε, χώρες που εδώ και 40-50 χρόνια ε, είχαν πόλεμο μεταξύ τους, είχαμε την Ευρώπη τη διαμάχης των πολέμων, ε, του μίσους όλα αυτά εξαφανίστηκαν χάρη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και αυτό φυσικά, όπως σας είπα, είναι αξιοζήλευτο. Και φαίνεται ότι εμείς, αυτοί που το βιώνουμε, δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η πρόκληση, διότι ήθελα να είμαι σύντομος και ολοκληρώνω με αυτό. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι διατεθειμένο να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα προεκλογική περίοδο, η οποία, όπως θα διαπιστώσετε όλοι, είναι διαφορετική κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχουμε πολλές πολιτικές φωνές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το κόμμα μου, οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι, ε, οι φιλελεύθεροι, να κάνουν μια συζήτηση που θα είναι ενημερωτική για όλους και διάφανη και θα μας επιτρέψει ολονών να διαμορφώσουμε άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο Σεμπάσιαν τώρα να μας διαβάσει λίγο τι γίνεται στο Twitter, ποιες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από το πάνελ εδώ. Έχουμε 130 δημοσιογράφους στην αίθουσα, φαντάζομαι ότι θα είναι πολλές οι ερωτήσεις. Έγινε πολλή συζήτηση, κυρίως για τα πιο ακραία κόμματα, τα οποία ε, αυξάνουν τα ποσοστά τους στην Ευρώπη, το Front National ε, στη Γαλλία που είναι πλέον το ε, μεγαλύτερο κόμμα στη Γαλλία από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, ε, η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Τα πιο ακραία κόμματα λοιπόν φαίνεται να λαμβάνουν πολύ ενδιαφέρον και υπήρχε και μία ερώτηση σε ποιο βαθμό οι ε, ευρωβουλευτές αντιλαμβάνονται σοβαρά αυτή τη διαμαρτυρία από πλευράς πολιτών. Θεωρούν ότι είναι απλώς ομάδες πίεσης και ελληπή ενημέρωση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Ποδηματά που είναι από την Ελλάδα και ξέρει περισσότερα για τη Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι μπορείτε να πείτε εσεί δύο λόγια. Επιτρέψτε μου, προς τιμή των Ελλήνων συναδέλφων που είναι στην αίθουσα, να μιλήσω κι εγώ τη μητρική μου γλώσσα. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, στις διαφορετικές της εκφάνσεις, γιατί στην ε, Ελλάδα το φαινόμενο της ε, ε, χρυσή αυγή είναι ένα φαινόμενο ενός μορφώματος που έχει ακραία φασιστικά, νεοναζιστικά χαρακτηριστικά. Είναι ένα φαινόμενο ωστόσο που μας απασχολεί πάρα πολύ στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο, και στο εθνικό επίπεδο ασφαλώς ε, να πω δύο κουβέντες για αυτό που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή για όσους συναδέλφους είναι εδώ και δεν τα παρακολουθούν από κοντά. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι πρόσφατα ε, μετά από μια σειρά ε, καταγγελίες που αφορούσαν στις δραστηριότητες στελεχών ακόμα και της ηγετικής ομάδας της χρυσή Αυγής με διαδοχικές ε, ε, βίες επιθέσεις, απόπειρες δολοφονίας ε, σε βάρος μεταναστών κυρίως, στη συνέχεια όμως επιθέσεις σε βάρος πολιτικών αντιπάλων και κορυφαίο βεβαίως από τρόπο γεγονός την ψυχρο δολοφονια δολοφονία ενός 34χρονου νέου ε, ράπερ. Στη συνέχεια όλων αυτών των γεγονότων ε, μαζεύτηκαν τα αναγκαία στοιχεία σε επίπεδο διοκτικών αρχών, υποβλήθηκαν οι φάκελοι στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη προχώρησε, ε, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, στη σύλληψη της μεγάλης πλειοψηφίας της ηγετικής ομάδας αυτής της οργάνωσης, η οποία είναι σήμερα προφυλακισμένη εν αναμονή της ε, διεξαγωγής μιας δίκης κάτω από πολύ βαριές κατηγορίες που αφορούν την ε, σύσταση και τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Γιατί είναι άλλο πράγμα ε, η ιδεολογία και οι πολιτικές θέσεις. Η δημοκρατία είναι πολύ ισχυρή για να είναι ανεκτική ακόμα και σε θέσεις που στην πραγματικότητα επαγγέλλονται ε, την, ε, τον περιορισμό της ή και την κατάλυσή της, αλλά δεν είναι και δεν μπορεί να είναι καθόλου μα καθόλου ανεκτική σε ό,τι αφορά πράξεις και συμπεριφορές που παραβιάζουν την ουσία του δημοκρατικού ε, πολιτεύματος σε όλα τα επίπεδα. Αυτά σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις στην Ελλάδα σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Όμως η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο και νομίζω ότι αυτό υπογραμμίστηκε και από τους ε, άλλους ε, ε, ομιλητές. Υπάρχει μία άνοδος της ακροδεξιάς, άνοδος εξτρεμιστικών κινημάτων και μορφωμάτων σε όλη την Ευρώπη, άνοδος του ευρωσκεπτικισμού και αυτό έχει να κάνει και με την κρίση και κυρίως με το είδος των απαντήσεων που έδωσε η Ευρώπη στη διάρκεια της κρίσης. Και όταν λέω το είδος των απαντήσεων, ε, εννοώ ότι οι πολίτες, και αυτό δεν αφορά μόνο τις χώρες του Νότου, που κυρίως πλήττονται, πλήγησαν από την κρίση, αφορά και τις, τους πολίτες ε, βορειοευρωπαϊκών και κεντροευρωπαϊκών χωρών, έχουν ε, την πεποίθηση την ε, βάσιμη πεποίθηση θα έλεγα ότι ε, αυτοί ήταν που σήκωσαν το μεγάλο βάρος αυτής της κρίσης. Οι πολίτες, οι φορολογούμενοι, στο νότο και στο βορρά, σήκωσαν το μεγάλο βάρος μιας κρίσης που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην αφετηρία της ήταν μια κρίση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ήταν μια κρίση λοιπόν που προκλήθηκε από την απειλή κατάρρευσης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σε πρώτη φάση η κινητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν για να διασωθούν οι τράπεζες και να αποφευθεί η συνολική κατάρρευση λόγω των εξαιρετικά καταστροφικών συνεπειών που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ε, με περικοπές αιματηρές στις χώρες του Νότου, ε, αλλά και με περιοριστικές πολιτικές στις χώρες του Βορρά, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι σήκωσαν και σηκώνουν το μεγάλο βάρος της κρίσης. Απέναντι σε αυτό διαμαρτύρονται. Ε, εγώ λέω λοιπόν ότι η διαμαρτυρία είναι θεμητή. Η διαμαρτυρία όμως, ε, όταν είναι μια διαμαρτυρία σκέτη που δεν περιλαμβάνει πρόταση, ε, ενέχει τον κίνδυνο να περιπλέξει το πρόβλημα αντί να, να ανοίξει μια, ε, ένα δρόμο για την, για την αντιμετώπιση του. Λέω ότι ε, πρώτα απ' όλα αυτό που υπογράμμισα και στην αρχή, ότι υπάρχει η ανάγκη για να διαμορφωθούν αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη αυτήν τη διάσταση που έλεγα πριν, της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα στα κράτη-μέλη και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης. Οι λύσεις θα πρέπει να είναι συνολικές. Οι λύσεις θα πρέπει να αναζητώνται στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο επίπεδο, αν μιλάμε για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και στο εθνικό επίπεδο ασφαλώς, αλλά το εθνικό επίπεδο από μόνο του δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Και το δεύτερο, και βάζω μία τελεία, ε, η, η διαμαρτυρία, ε, η ακραία διαμαρτυρία μερικές φορές, η απόρριψη, η ισοπεδωτική απόρριψη του κατεστημένου, του υπάρχοντος συστήματος, όταν οδηγεί ε, στην ανάσυρση επιλογών που έχουν δοκιμαστεί στην ιστορία, έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν. Ο φασισμός και ο νεοζισμός ε, έχει ε, ε, αφήσει τεράστιες πληγές στην Ευρώπη. Λοιπόν, άρα λέω ότι οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών έχουν πολύ μεγάλη δύναμη στην πραγματικότητα να αλλάξουν τα πράγματα. Πιστεύω πάρα πολύ, σε αυτό δεν ξέρω, είσαστε και πολύ νεότεροι, το τραγούδι της Patti Smith «People have the power». I am very much convinced Uh, um, Είμαι βέβαιη ότι έτσι είναι. Οι άνθρωποι έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Αλλά νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο ότι όντως έχουν την εξουσία στα χέρια τους και μπορούν αυτοί να αλλάξουν το ρουν σε εθνικό επίπεδο, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο της ιστορίας πριν από τις ευρωεκλογέ, οι οποίες αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικές, διότι και το πλαίσιο της κρίσης αλλάζει τα πράγματα, αλλά και γιατί πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα άμεσα να εκλέξουμε το νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς έχουμε την εξουσία στα χέρια μας, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εξουσία και να προτείνουμε κάποια πράγματα και όχι απλώς να διαμαρτυρόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε. But before you ήσασταν κι εσείς ε, δημοσιογράφος πριν από χρόνια και η κυρία <clears throat> η είπε ότι στην Πορτογαλία ο κόσμος μισεί τώρα τους πολιτικούς. Αυτό πώς σας κάνει να αισθάνεστε. Ήσασταν και εσείς δημοσιογράφος εσείς, είστε τώρα από την άλλη πλευρά. Τι νιώθετε, σας κατηγορούν, ε, τι, τι, τι λύσεις μπορείτε να δώσετε σε καιρού απελπισίας. Ε, people ναι, ο κόσμος κατηγορεί τους πολιτικούς και διαμαρτύρεται. Τώρα όμως ε, περισσότερο ως δημοσιογράφος για 22 χρόνια και όχι ως πολιτικός, εγώ υποστηρίζω προσεγγίσεις που να είναι, πώς να το πω, δεν πρέπει να βλέπουμε τους πολιτικούς ως σύνολο και να λέμε ότι είμαστε υπέρ κατά της γενικής τάσης. Αυτό είναι εις βάρος όχι για τους των πολιτικών, όχι των θεσμών, είναι εις βάρος των ίδιων των πολιτών. Νομίζω πως πρέπει να προσπαθήσουμε να όρθολο, να δώσουμε μια έννοια, μια λογική στα όσα συμβαίνουν, ποια ήταν τα αίτια της κρίσης και ποιες είναι οι σωστές επιλογές για να προχωρήσουμε. Το να απορρίπτει κανείς τους πολιτικούς συλλήβδιν και την πολιτική δεν είναι η λύση, γιατί αυτό δίνει βάση και χώρο για τους ε, εξτρεμισμούς, για τις ακρότητες, για τα ακροδεξιά κόμματα. Δεν είναι λύση αυτή. Είναι πραγματικά κίνδυνος και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πιο περίπλοκη κατάσταση από αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω τον ε, κύριο Χαφ από το Λίβερπουλ και την, ε, το, κόμμα της ανεξαρτησίας ασχοληθήκατε με το ε, νεότητα του κόμματος ανεξαρτησίας πριν να ακούσουμε άλλες ερωτήσεις, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τα σχόλιά σας για αυτό το θέμα, που είναι βέβαια ο αντίκτυπος των νέων κοινωνικών κινημάτων στα πολιτικά κόμματα, καθώς προχωρούμε προς τις επόμενες ευρωεκλογέ. Είναι πρόβλημα το γεγονός ότι υπάρχει κίνημα, κίνηση προς την ε, ακραία τις ακρότητες. Ε, το είδαμε με την ε, στήριξη του ε, Front National στη Γαλλία και σίγουρα στην Ελλάδα με την ανάδεση της χρυσή αυγή. Πιστεύω ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ίδιες οδηγούν τον κόσμο και κυρίως τους νέους στις αγκάλες των εξτρεμιστικών κομμάτων. Δείτε και τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχουμε την αφαίρεση στην ουσία της δημοκρατίας, την κατάργηση των δημοκρατικά εκλεγμένων ε, ε, ε, πολιτικών και στη θέση αυτών έχουμε μια τρόικα η οποία υπαγορεύει την οικονομική πολιτική της Ελλάδας και έχουμε αυτή τη στιγμή 50% ανεργία στην Ελλάδα. Δηλαδή μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων οι οποίοι ριζοσπαστικοποιούνται. Στην ε, Ισπανία είμαστε στο 35%. Άλλο ε, πρόβλημα είναι ότι έχουμε από εκεί διαρροή των εγκεφάλων. Ο κόσμος ε, φεύγει πάνε στη Γερμανία, πάνε στη Νότια Αμερική όπου μπορούν. Όταν ο κόσμος απελπίζεται, προτείνει να πηγαίνει στα άκρα. Στα άκρα. Και το πρόβλημα για την Ισπανία και την Ελλάδα ιδιαίτερα είναι ότι είναι παγιδευμένοι σε μια πολιτική στην οποία δεν θα έπρεπε να είναι παγιδευμένοι. Αν θέλουν να κινηθούν οι οικονομίες τους και θέλουν να δώσουν μια όθεση, μα δεν μπορούν να συνεχίζουν με αυτή την κατάσταση με τα επιτόκια και τα... Ε, που, που δεν βοηθούν την οικονομία. Το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να επιτρέψει στην Ελλάδα να φύγει από το ευρώ. Στη χώρα μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε 22% ανεργία των νέων. Πρόκειται για ένα εκατομμύριο παιδιά ανάμεσα στα 18 και τα 24 που δεν μπορούν να βρουν δουλειά είναι, κακό, είναι βέβαια κακό, αλλά και δόξα σε Θεό δεν είναι τόσο χάλια όσο στην Ισπανία και στην ε, Ελλάδα. Και δόξα σε Θεός που δεν μπήκαμε στο ευρώ όταν ήθελε το εργατικό κόμμα να μας βάλει. Γιατί εμείς έχουμε έλεγχο του και νομίσματό μας, δεν είμαστε παγιδευμένοι σε ένα νόμισμα το οποίο έχει φτιαχτεί για να βολεύει τη Γερμανία. Το πρόβλημα που έχουμε όμως εμείς ε, και είναι αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα στην ε, Αγγλία και είναι ο λόγος για τον οποίο ο κόσμος μας δεν μπορεί να βρει δουλειά είναι γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει την ε, πολιτική μετανάστευση ιδιαίτερα από την Ανατολική Ευρώπη. Όταν επιτρέψαμε να ανοίξουν τα σύνορά μας το 2004 σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη η εργατική κυβέρνηση είπε πως μόνο 13.000 κόσμος θα έρχονταν. 200.000 ήρθαν τον πρώτο χρόνο, μόνο τον πρώτο χρόνο. Και από τότε έχουν έρθει άλλα δύο εκατομμύρια. Και το πρόβλημα είναι ότι αν πας οποιαδήποτε πόλη, στη Κομόπολη, μπαράκι, εστιατόριο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ακούς αγγλικά, δεν δουλεύει κανένας εγγλέζος. Κυρίως Ανατολικοευρωπαίοι. Και δεν τους κατηγορώ που ήρθαν, ε, γιατί κατά σε πολύ μεγάλο βαθμό βελτιώνουν τους μισθούς τους. Αλλά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την Ένωση και την κυβέρνησή μας. Γιατί αν θέλει κανείς να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων στη Βρετανία, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την μετανάστευση. Γιατί τα δύο αυτά πάνε χέρι-χέρι. Ένας από τους λόγους για τους οποίους είδαμε την ανεργία να αυξάνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ανάπτυξη των, ευρω... των ευρωσκεπτικιστών είναι γιατί δεν μπορούμε να, να αντιμετωπίσουμε το θέμα της μετανάστευσης. Και ο κόσμος, οι νέοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά γιατί η αγορά έχει κορεστεί. Φανταστείτε τι θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου που θα αρχίσουν να έρχονται και οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι. Άλλα 30 εκατομμύρια κόσμος που θα μπορεί ωραιότατα να έρθει. 50.000 άνθρωποι τον χρόνο υπολογίζεται ότι θα έρθουν για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ήδη οι νέοι δεν έχουν δουλειά. Άμα έρθουν κι άλλοι, ε, ο κόσμος θα αρχίσει να πικραίνεται, θα αρχίσει να θυμώνει. Ήδη κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, δείχνουν πως η πλειοψηφία των Βρετανών αυτή τη στιγμή θα ψήφιζαν να φύγουμε από την Ένωση. Η μεγάλη πλειοψηφία των Βρετανών θέλουν δημοψήφισμα και γι' αυτό και ο Κάμερον έδωσε αυτή την υπόσχεση για δημοψήφισμα για το 2017. Το πρόβλημα που έχουμε λοιπόν είναι στα, στα κράτη της Νότιας Μεσογείου, είναι παγιδευμένα σε ένα νόμισμα στο οποίο δεν θα έπρεπε να είναι, ιδιαίτερα στην Ελλάδα εκλεγμένος κόσμος που διευθύνει υποτίθεται την, την, ε, την οικονομία και οδηγεί τους νέους στις αγκαλιές των ε, ριζοσπαστικών κομμάτων. Στη χώρα μου είναι ότι ενώ, το πρόβλημα ότι ενώ είμαστε μέλη της Ένωσης ε, δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα σύνορά μας και δεν μπορούμε να πούμε ποιος θα μπαίνει και ποιος θα βγαίνει από τη χώρα μας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα είναι το βασικό θέμα στις ευρωεκλογές του χρόνου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Φανταστικό να έχουμε τόσο μεγάλη ποικιλία απόψεων. Έχετε το λόγο για ερωτήσεις. Και μετά έχω τον κύριο με τα γελιά και το μαύρο που κάμισο. Εντάξει, παρακαλώ να μας συστηθείτε. Γεια σας, ονομάζομαι Μάριον Μπάχερ και εργάζομαι για την Αυστριακή Ραδιοτηλεόραση και σε σχέση με, με την μετανάστευση θέλω να ρωτήσω τι επιπτώσεις έχει η μετανάστευση στα κοινωνικά κινήματα γιατί αν πολλοί κόσμος φεύγει από τον Νότο και πάει προς το Βορρά ή προς τη Βραζιλία, την Αφρική όπως γίνεται πούμε με την Πορτογαλία επηρεάζει αυτό τα κοινωνικά κινήματα και άλλη πλευρά είναι επηρεάζει την ε, συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Γιατί, για παράδειγμα, όταν ο κόσμος εργάζεται στην Ελλάδα, μάλλον Έλληνες που εργάζονται στη Γερμανία, ή Πορτογάλοι, ή Ισπανοί, ίσως να μην θέλουν να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Πώς μπορούν εκείνοι να σημάνουν την αλλαγή για την ίδια τους τη χώρα, ας πούμε. Ευχαριστώ. Και εσείς με τα γελιά. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Μάρκα Σερένα από τη Βαρκελόνη. Όπως ξέρετε και οι συνάδελφοι εδώ, εμείς ε, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος ε, μας μιλά, το πιο σημαντικό είναι, από αυτά που μας λένε είναι αυτά που δεν μας λένε. Και γι' αυτό και πραγματικά εντυπωσιάζομαι με τον κύριο από την Ισπανία εδώ, γιατί σήμερα μιλάμε για τα κοινωνικά κινήματα και μιλάμε για τα εθνικά προβλήματα και τις ευρωπαϊκές λύσεις. Και όπως γνωρίζετε, ακόμα και αν μίλησε για την Αραβική Άνοιξη, έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά κινήματα στην Καταλωνία. Είχαμε μια διαδήλωση όπου συμμετείχε 1,5 εκατομμύριο κόσμος πέρυσι. Πρόσφατα άλλη διαδήλωση με ένα εκατομμύριο κόσμο που κρατούσαν τα χέρια τους. Γίνεται πολλής λόγος για εξτρεμισμό, για κοινωνικά κινήματα, για, ε, ραντικα, ε, για ριζοσπαστικά κινήματα. Το θέμα είναι πάντως πως το 71% των ανθρώπων που ζουν στην Καταλωνία ζητούν δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο κόσμος αν θέλει να είναι μέρος της Ισπανίας ή όχι. Και μόνο 21% του πληθυσμού λέει ότι δεν θέλει να ψηφίσει. Και ακόμα και έτσι είμαστε μπλοκαρισμένοι. Διότι το κόμμα που αντιπροσωπεύει ο κύριος Ευρωβουλευτής μπλοκάρει την κατάσταση στην Ισπανία αλλά και εδώ στην Ευρώπη. Το ερώτημά μου είναι τι να περιμένουμε από την Ευρώπη. Αφού βλέπουμε ότι 71% του κόσμου ζητά δημοψήφισμα και δεν τους απευθύνουν. Γιατί λέει δεν μπορείτε να ψηφίσετε. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Τι να περιμένουμε τότε από την Ευρώπη. Η Ευρώπη για την ώρα πει την ίσα, δεν εκφράζει την άποψή της και λέει ότι δεν είναι δικό της θέμα. Ωραία. Άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Οι τρεις επόμενοι και λίγο σύντομοι γιατί μας τελειώνει ο χρόνος. Edgar Mannheimer από το UFPF Learn στη Σουηδία, ραδιοφωνικό σταθμός. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η ιδέα ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ανεργίας των νέων και του εκθρεμισμού. Και στη Σουηδία και στην Νορβηγία, για παράδειγμα, η οικονομία πηγαίνει μάλλον καλά παρά την κρίση και εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλη υποστήριξη λαϊκιστικών κομμάτων κατά των μετανιστών. Και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα. κατά πόσον θεωρείτε εσεί ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ εκκρεμισμού και εξτρεμισμού και ανεργία. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ ο συνάδελφος ξεκίνησε την ερώτηση, αλλά δεν τελείωσε, αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε για τα κοινωνικά κινήματα στην Ισπανία. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι προς τον ε, κύριο Αντιρόνιο Λόπεθ ε, Ιστουρίθ. Πώς βλέπετε λοιπόν εσείς τα κινήματα τα οποία στην Ισπανία ήταν πολύ μεγάλα και ε, είχαν τόσο μεγάλη παρουσία. Πώς θα εξηγείτε σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και τι σχέση θεωρείτε ότι έχουν με την Αραβική ε, ε, άνοιξη και το κίνημα Occupy. Συγγνώμη, από πού είστε? Γκρίνα Μπόλτ από τη Βιέννη και γράφω μια διατριβή για την κατάσταση στην Ισπανία και δεν αναφερθήκατε καθόλου στο κίνημα αυτό. Καλό είναι να έχουμε κάποιες πληροφορίες. Η κυρία με το πράσινο μπλουζάκι. η ερώτησή μου και πάλι και για μένα για τον κύριο Λόπεθ. Ε, λέγομαι Μουνιώθ, είμαι από την Ισπανία. Η διαρροή εγκεφάλων είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ακόμα για την Ισπανία. Πώς θα διαβιβάσουμε το μήνυμα σε όλους αυτούς τους νέους που είναι επιφυλακτικοί διότι χρειάστηκαν να μεταναστεύσουν προκειμένου να αποκτήσουν ένα καλύτερο μέλλον. τους λέμε, πώς θα τους πείσουμε ότι αυτοί έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Διότι είναι πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Ε, πώς μπορεί να αλλάξει το... τα πράγματα, πώς μπορούν οι νέοι να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Καλημέρα σας. Ειλίν από την Ιρλανδία. Αναφέρεστε στη μετανάστευση των νέων και την ανεργία των νέων, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει όσα πρέπει προκειμένου να επικεντρωθεί στην επιχειρηματικότητα των νέων. Ναι, πολύ καλή παρατήρηση. Άλλες ερωτήσεις? Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με τον Πολ και μετά να δώσουμε το λόγο σε όλους με τη σειρά από 2-3 λεπτά. Θα απαντήσω στη σουηδική ερώτηση, αν υπάρχει σχέση μεταξύ εκκρεμισμού και μετανάστευσης εξτρεμισμού και ανεργίας. Κυρίως ανεργία και εξτρεμισμός. Η ιστορία της Ευρώπης σας διδάσκει ότι όντως ισχύει αυτό. Όταν ο κόσμος είναι άνεργος, δεν έχει χρήματα, ε, είναι χωρίς ελπίδα, τότε οδηγούνται προς τον εξτρεμισμό όπως ε, ε, πάει η πεταλούδα στο φως. Ε, είναι αυτή η αίσθηση ότι δεν ανήκουν πουθενά, ε, η απελπισία και τελικώς νιώθουν ότι η μόνη διέξοδος είναι να στραφούν σε εξτρεμιστικά κινήματα. Και αυτό ξεκινάει με διαδολώσεις στους δρόμους. Ε, όταν μιλάω για ακραία κινήματα αναφέρομαι είτε σε ακραριστερά είτε σε ακραδεξιά για την Καταλωνία. Ως πρώην κάτοικος της Βαρκελόνης και εγώ ε, να σας πω ότι ναι μεν ε, κατανοώ τους ε, Καταλανούς αλλά δεν μπορείτε να περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σας υποστηρίξει για το δημοψήφισμα. Ήμουνα σε μια συνέντευξη τύπου πριν από κάνα δύο χρόνια όπου ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο ανέφερε ότι τα ε, δημοψηφίσματα είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Δυσάρεστη κατάσταση αντιλαμβάνεστε. Αυτό λοιπόν σημαίνει συμβαίνει με το δημοψήφισμα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σας δώσει ε, τα ο, πράσινο φως για το τι να κάνετε, να ακολουθήσετε το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς δώσαμε τη δυνατότητα στη Σκωτία να κάνει δημοψήφισμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διαφορά ε, για την Καταλωνία ή τη Σκωτία. Η διαφορά είναι ότι η Σκωτία είναι η πιο ε, βόρεια άκρη ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά πάσα πιθανότητα, του Ηνωμένου Βασιλείου συγγνώμη, και κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσει να μείνει γιατί θα είναι μόνη της αλλιώς στην άκρη, ενώ η Καταλωνία είναι με στη μέση. Ένας λόγος για τον οποίο στο Ηνωμένο Βασίλειο είμαστε υπέρ του δημοψηφίσματος είναι γιατί όταν ενταχθήκαμε στην τότε ΕΟΚ το 1975 μέσω δημοψηφίσματος, δεν μπήκαμε, ψηφίσαμε αν θα πρέπει να μείνουμε ή να ε, φύγουμε, τότε ψηφίσαμε για το εμπόριο και ε, την οργάνωση αυτών των σχέσεων. Η ΑΟΚ του 1975 δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα. Ούτε συζητούσαμε σημαίες, ούτε κοινοβίλια, ούτε ανοιχτές πόρτες για τη μετανάστευση. Συζητούσαμε εμπόριο, εμπορικές σχέσει. Και αν ε, ήσασταν 24 ετών σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ψηφίσατε ποτέ για το αν θα πρέπει να ημείνουμε ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε εγώ δεν είχα γεννηθεί καν. Και ένας από τους λόγους ε, από τους ανθρώπους που, δεν που υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, έρχονται στο κόρμα μου ε, είναι γιατί πραγματικά θεωρούν ότι δεν τους έχει ρωτήσει κανείς και νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Ισπανία. Δεν ξέρω τι γλώσσα πρέπει να μιλήσω, μάλλον Ισπανικά πρέπει να απαντήσω. Διότι αναφέρεστε συνέχεια στην Ισπανία και στην Καταλωνία εδώ και νομίζω ότι μπορώ να δώσω τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, από λίγο πιο μακριά, από την Πράγα, από την Τσεχία. Διότι εδώ ρωτάμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνουν οι πολιτικοί για την Καταλωνία και την Ισπανία. Η απάντησή μου είναι ότι εγώ δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε μάλλον. Και αυτή είναι η ερώτηση, διότι εμείς αρχίζουμε να μιλάμε, εγώ άρχισα να μιλάω για την επανάσταση και την εξέλιξη. Και σας είπα και το τρίτο, την ταχύτητα και οι συνάδελφοι το σχολίασαν και αυτοί. Η ταχύτητα η οποία αυξάνεται συνεχώς ε, στην πολιτική του σήμερα. Αν δούμε τι γινόταν πριν από 10 μόλις χρόνια, η πολιτική γινόταν με μάχες και στους δρόμους. Ε, πριν από 60-70 χρόνια η πολιτική ήταν σαν το θέατρο περίπου. Δηλαδή, υπήρχε ένα βήμα στο οποίο ήταν ε, οι ε, παράγοντες, οι ηθοποιοί, οι επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων και ο κόσμος κοιτούσε και μπορούσε απλώς να συμμετέχει με την ψήφα του. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δέκα χρόνια, και αυτό είναι η ταχύτητα, άλλαξε πάρα πολύ η πολιτική. Εμείς δεν είμαστε πλέον αυτοί που αποφασίζουμε. Ξαφνικά σηκώνεστε εσείς, εσείς ε, θα έχετε το τέλειο tweet, θα σας κάνουν retweet 10 εκατομμύρια άνθρωποι και έτσι γίνεται η πολιτική σήμερα. Και το ερώτημα είναι, είναι καλό ή κακό αυτό, διότι αν θέλουμε να κάνουμε βιώσιμη πολιτική, χρειαζόμαστε χρόνο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συνένεση, να μην κάνουμε ακραία πράγματα. Η απάντησή μου λοιπόν είναι απλή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Καταλωνία και την Ισπανία. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω ε, είναι ότι στη χώρα μου, στην Τσεχική Δημοκρατία, προσφάτως έχουμε αρκετούς Ισπανούς που έρχονται να εργαστούν στη χώρα και εγώ το θεωρώ θετικό, διότι πολλοί μαθαίνουν Τσέχικα που είναι μια γλώσσα η οποία είναι μειονοτική αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ σας ευχαριστώ και να συνεχίσουμε στα Ισπανικά. You said um, first about the extremes. We're very worried. Να σας πω καταρχάς ότι για τα εξτραμιστικά κινήματα μας ανησυχούν πολύ. Είναι κινήματα τα οποία ε, δυστυχώς δεν είναι δημοκρατικά. Εγώ έχω την εμπειρία ακροαριστερών ανεξάρτητων κινημάτων στην Ισπανία που οδήγησαν στην ΕΤΑ, την οργάνωση των Βάσκων Αστυνομιστών. Και όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν μόνο δημοκρατικά και μόνο ενωμένοι. Εμείς, οι σοσιαλιστές, ε, οι ε, μετριοπαθείς οι εθνικιστές, οι οποίοι δεν συμμερίζονται την ίδια άποψη και θέλουν να συμμετέχουν στη δημοκρατία, όλοι μαζί καταφέραμε να λύσουμε αυτό το θέμα και αυτή είναι η δύναμη της Ισπανίας. Και έτσι θα πρέπει να είναι και στην Ελλάδα. Όλες οι πολιτικές ομάδες ενωμένες κατά της χρυσή αυγή και αυτού που αντιπροσωπεύει. Εάν δουν ότι υπάρχουν διαμάχες μεταξύ των δημοκρατικών δυνάμεων, τότε θα αρπάξουν την ευκαιρία και τότε εσείς ε, δεν θα μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα. Πάντα η δημοκρατία είναι η λύση. Παρακολουθούμε βέβαια στενά το φαινόμενο αυτά και θέλω να τα καταδικάσω, να καταδικάσω τη δολοφονία αυτού του νέου ανθρώπου. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε αλλού. Δυστυχώς στην Ισπανία έχουμε πικρά πείρα του φασισμού και των, ε, της ακροδεξιάς και φυσικά είναι ε, άσχημες οι αναμνήσεις. Κάποιοι από εσά έθεσαν ε, μια ερώτηση για τη μετανάστευση. Εγώ έχω μια αρχή. Δεν μπορεί να φέρνεις ανθρώπους να σε βοηθήσουν όταν έχει τα μέσα και μετά να τους απολύει όταν δεν έχεις πλέον τα μέσα να τους πληρώνεις. Αυτό δεν είναι στην ανθρώπινη φύση. Αυτό έγινε γιατί ε, ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι γιατί τους χρειαζόμασταν. Μας βοήθησαν στην ώρα ανάγκη και τώρα ξαφνικά αλλάζουμε στάση και θέλουμε να του πετάξουμε όλου έξω. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Έπρεπε να ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στο παρελθόν ίσω. αλλά τώρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να του πετάξουμε όλου έξω από την πόρτα. Πρέπει να υπάρχει σαφή και διάφανη πολιτική. Υπάρχει και ο ανθρώπινο παράγοντα εδώ. Την ερώτηση για όλους αυτούς τους Ισπανούς που πάνε σε άλλες χώρες για να εργαστούν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Ισπανική κυβέρνηση ώστε να επιστρέψουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν γιατί αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες. Αυτό είναι λογικό. Και η Ισπανία δυστυχώς δεν είναι η πρώτη περίπτωση για όσους ε, θυμούνται λίγο τα πράγματα. Ήταν χώρα μετανάστευση και στο παρελθόν και έγιναν δεκτοί οι Ισπανοί και στη δεκαετία του 60 και του 70 σε άλλες χώρες. Δεν είναι αυτό που θέλουμε και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εργάζεται ώστε να μετριάσει λίγο τις συνέπειες. Τώρα, το κίνημα Τη 15 Μαρτίου. Εγώ συμμετέχω σε μια γενιά πολιτικών που παρακολουθεί πολύ στενά ποια είναι τα αιτήματα του κινήματος 15 ε, μη. Σήμερα δεν είναι τα ίδια τα πράγματα όπως πριν από δύο χρόνια. Νομίζω ότι εξελίχθηκε ε, το οικονομικό τοπίο, υπάρχουν κάποιες ελπίδες, αλλά δεν έχουν τελειώσει όλα. Uh, Τίποτα δεν έχει λυθεί και ακόμα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε και στις ε, απαιτήσει ε, σε κοινωνικό επίπεδο των νέων. Εγώ πάντα σεβάστηκα το τμήμα του 15μη που δεν ήταν πολιτικοποιημένο, ήταν ένα αυθόρμητο ε, κίνημα διαμαρτυρίας νέων. Αυτό έτυχε του αμόριστου σεβασμού μου. Αλλά η πολιτική παρέμβαση που ήρθε στη συνέχεια δεν ήταν το ίδιο. Όσον αφορά τώρα το θέμα της Καταλωνίας και τη σχετική ερώτηση, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αυτό που δεν είπατε είναι ότι υπήρξε και μια διαδήλωση το περασμένο Σαββατοκύριακο από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν η Καταλωνία να ανήκει στην Ισπανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ισπανία. Έχουμε και την άλλη πλευρά. Ε, δεν το είπα γιατί εγώ αναφέρομαι στην Ευρώπη βέβαια, αλλά η ανησυχία μου δεν είναι ο εθνικισμός ε, ο εθνικισμός οδήγησε σε χρόνια πολέμων στην Ευρώπη. Για μένα η απάντηση είναι Ευρώπη. Η απάντηση για την Καταλωνία και την Ισπανία είναι Ευρώπη. Το 70% του ισπανικού λαού νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου. Εάν και εφόσον λοιπόν υπήρχε δημοψήφισμα, θα έπρεπε να γίνει σε όλη την Ισπανία, γιατί και αυτοί έχουν δικαίωμα να μας πούν την άποψή τους. Διότι είμαστε συνταγματικό κράτος, δημοκρατικό και η, οποία, η, γνώμη των 47 εκατομμυρίων Ισπανών έχει κάποια βαρύτητα. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε στην απέξω σε περίπτωση που υπάρξει δημοψήφισμα. Εχθές ή σήμερα νομίζω διάβασα ε, στις εφημερίδες ότι 9 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτό το οποίο ζητάει η αυτόνομη περιφέρεια της ε, ε, Καταλωνίας σε αυτή τη συζήτηση για τον προπολογισμό που γίνεται τώρα και είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας που δίνει μάχη για το δημοσιονομικό έλλειμμα όχι μόνο στην Ισπανία, γιατί στην Καταλωνία, γιατί η Καταλωνία χρωστάει 50 δισεκατομμύρια ευρώ η Ισπανία λοιπόν θα βοηθήσει την Καταλωνία, τη Γαλλικία, τη χώρα των Βάσκων θα δώσουμε μια μάχη μαζί. Και... Στο λαό μας, στην Καταλωνία, στη χώρα των Βάσκων, στην Καστήλη θα φέρουμε πάλι πίσω το δικαίωμα στην ευημερία, την ανεργία και όλα τα δικαιώματα τα οποία έχασα. Πάντα ρωτιέμαι γιατί όλα αυτά τα κινήματα, συγγνώμη γιατί είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις, δεν ξέρω αν θυμάστε την τελευταία φορά ε, με τους Γερμανούς, ε, τέθηκαν όλες αυτές οι ερωτήσεις, πρέπει να απαντήσω. Μακάρι να χρειαζόταν να μιλήσω μόνο για την Ευρώπη, αλλά αυτά με ρωτήσατε και πρέπει να απαντήσω σε αυτά που με ρωτήσατε. Είναι καθήκον μου. Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω και δεν ξεχνώ και τίποτα. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι όπως και ο Έντβαρτ, όταν γνωρίζω πολύ καλά μια κατάσταση, μπορεί κάποιος να σας θέλει να σας πει ότι είμαι φασιστής από το Παρτίδο Ποπουλάρ, που δεν θέλω να ακούγεται η γνώμη των ανθρώπων. Όχι, εγώ είμαι από τη Μαγιόρκα, ε, μιλάω καταλανικά ε, και ε, καταλαβαίνω πολύ καλά την κατάσταση. Και Ήμουν από τους πρώτους που ήμουν υπέρ του δικαιώματος της γλώσσας της Καταλων... στην Καταλωνία, στη Μαγιόρκα. Και η αυτονομία στην Καταλωνία, ο βαθμός αυτονομίας που έχει η Καταλωνία, η χώρα των Βάσκων, η Γαλλικία, είναι μεγαλύτερη από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Είναι περισσότερη από ό,τι στη Φλάνδρα εδώ στο Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, περισσότερη από οπουδήποτε αλλού. Ε, στην αρχή δεν υπήρχαν αρκετές γνώσεις για το τι ε, συνέβαινε στην Ισπανία. Και επειδή εγώ είμαι προϊόν αυτού του αυτόνομου συνταγματικού κράτους ε, στην Ισπανία, χρειάστηκε να το εξηγήσω πολλές φορές και εντός ε, του ΕΛΚ. Όλοι, για παράδειγμα, στο ΕΛΚ γνωρίζουν ότι είμαι πολύ καλός φίλος της Ουγγρικής μειονότητας στη Ρουμανία. Πάντα προασπίζουμε αυτές τις μειονότητες διότι εντός του συνταγματικού κράτους της Ρουμανίας υπάρχει μια ουγγρική μειονότητα που δίνει μάχη για τη γλώσσα της, για την περιοχή τους και πάντα εγώ είμαι υπέρ αυτών των μειονοτήτων. Πιστεύω σε αυτή τη μορφή της δημοκρατίας και θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση για τα 9 δισεκατομμύρια και για πολλά άλλα πράγματα και νομίζω ότι είναι καλό το γεγονός ότι η Ισπανία συζητά με τον πρόεδρο της Αυτόνομης Περιφέρειας της ε, Καταλωνίας και θα συζητεί, συνεχιστούν οι συζητήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Γνωρίζετε από τον τύπο ότι γίνονται συζητήσεις. Πάντα είναι εν εξελίξη συζητήσεις και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα καλό στοιχείο της ισπανικής πολιτικής. Να δώσω τώρα το λόγο στις κυρίες, ε, στην άλλη πλευρά του ε, πολιτικού φάσματος. Η κυρία Ζιν Λάμπερτ. Για την Καταλωνία δεν θα ακούσετε τίποτα το ιδιαίτερο από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. έχετε δίκιο ότι θεωρείται εθνικό θέμα, γιατί αν αρχίσει κανείς να λάβει θέση, να λαμβάνει θέση για μια χώρα, θα πρέπει να το κάνει για, για όλες τις χώρες. Για το δημοψήφισμα της Σκοτίας να είμαστε σαφείς ότι αυτοί οι οποίοι γούντε του Εθνικιστικού Κόμματος της Σκοτίας, υπερασπίζονται την Σκοτία εντός της Ευρώπης και γι' αυτό υπάρχουν αρκετά βρετανικά κόμματα που καθόλου δεν τους αρέσει η ανεξαρτησία της Σκοτίας. Για την επιχειρηματικότητα των νέων στα κονδύλια που έχουμε υπάρχουν κάποια κονδύλια για διάφορου τομεί τη επιχειρηματικότητα, τις μικροπιστώσεις και υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε σε σχέση με το τι θα ζητήσει η χώρα σας. Τα χρήματα υπάρχουν. Ε, βάλτε ε, τον νέους να τα ζητήσουν. Ε, τώρα, ε, υπάρχουν κάποιες χώρες όπου αν δει κανείς τα στοιχεία, τα κόμματα, τα ε, κρέα, τα πήγαιναν πολύ καλά και όταν πήγαινε καλά η οικονομία και πάνε χειρότερα τώρα που η οικονομία είναι λιγότερο καλά και αυξάνεται η ενεργεία. Δεν είναι άμεση η σχέση. Σίγουρα όχι όσον αφορά τις ακροδεξιές ε, παρατάξεις. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Έχουν να κάνουν με τις ανησυχίες του κόσμου για την παγκοσμιοποίηση, απώλεια ταυτότητας ε, και για κάποιους είναι και η απώλεια στάτους και εξουσίας μέσα στην κοινωνία. Είναι ένα, ένα πλέγμα αιτίων. Και όσον αφορά τώρα τα κοινωνικά κινήματα, ο κόσμος που κινείται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυνατότητα ψήφου σε τοπικό επίπεδο στη χώρα που διαμένει και, ψήφο, και δικαίωμα ψήφου για τι ευρωεκλογέ στη χώρα που διαμένει. Αλλά η online εκστρατεία και η σύνδεση δίνει τη δυνατότητα ε, ο κόσμος να εκφραστεί και να βοηθήσει, βοηθά να αναπτυχθεί η συζήτηση γιατί έτσι έχει μια ευρύτερη εμπειρία που μπορεί να συγκρίνεις πράγματα. Και ξέρουμε ότι Υπάρχει χώρος για βελτιώσεις, αλλά αυτό που είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι έχουμε δικαιώματα όταν, κινούμεθα, όταν μετακινούμεθα μέσα στην Ένωση. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όταν κινούμεθα, όσον κινούμαστε ε, και θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ενώσον υπάρχουν. Υπάρχει κίνημα αυτή τη στιγμή από διάφορα πολιτικά κόμματα και σε ορισμένε χώρε. για να περιοριστούν τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και τα δικαιώματα που έχει κανείς καθώς κυκλοφορεί στην Ένωση και θα πρέπει να είναι θέμα στις ευρωεκλογέ. Η προστασία δηλαδή των δικαιωμάτων των ανθρώπων που κινούνται, μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια από τις αξίες ε, δεν θα πρέπει δηλαδή να περιορίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του κόσμου προς το συμφέρον στενών εθνικών συμφερόντων. Κυρία ε, Ζουμπερ τώρα. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. <laughs> Κράτα. Το θέμα του εξτρεμισμού. Μιλήσαμε για εξτρεμισμό. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι θα πει εξτρεμισμός. Γιατί εάν μιλάμε για ανθρώπινα κινήματα που θεωρούν ότι άνθρωποι κάποιων χώρα είναι κατώτεροι και άλλοι πρέπει να έχουν δικαιώματα και άλλοι όχι, ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν είναι κινήματα ε, ανθρώπινα τα οποία πρέπει να ε, επιτρέπονται και να μην συγχέονται με κινήματα που θεωρούν ότι ότι το μοντέλο ανάπτυξης είναι οι ε, διαφορές στις αμοιβέ, οι διαφορές στα δικαιώματα. Δηλαδή δεν είναι όλα όσα είναι κόντρα στο σύστημα απαγορεύστεα, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει δυνατότητα να σκεφτεί κανείς κάτι διαφορετικό και να δημιουργήσει και να οικοδομήσει κάτι το οποίο είναι ένα διαφορετικό. Το θέμα της ακροδεξιάς, της ανάδεσης της ακροδεξιάς έχει να κάνει ακριβώς με το θέμα των ανισοτήτων. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχει δηλαδή πλούτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χώρα έχει το δικό της πλούτο, αλλά είναι άνισα κατανεμημένος ο πλούτος αυτός. Γιατί λοιπόν ε, όταν, δημιουργείται, όταν καταστρέφονται θέσεις απασχόλησης και δημιουργείται μεγαλύτερη ανεργία, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι ορισμένες ομάδες ε, οικονομικές και ορισμένες χώρες συγκεντρώνουν περισσότερο πλούτο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να διατηρηθούν οι ε, όμιλοι αυτοί οικονομικοί, να συσσωρεύσουν περισσότερο πλούτο και η διαδικασία κατάργησης και καταστροφής θέσεων απασχόλησης βοηθά στη δημιουργία αυτού του πλούτου και μάλιστα γίνεται μεταφορά των πόρων των εργαζομένων προς τους ε, οικονομικούς ομίλους. Αυτό βλέπουμε, αυτό διαπιστώνουμε. το το συμμετέχει σε κινήματα κόσμος ε, επειδή βλέπει να συμβαίνει αυτό, γιατί το να καταστρέφουμε τις ζωές του κόσμου δεν χρησιμεύει σε τίποτα και βλέπουμε ότι αυτός είναι, μας παρουσιάζουν ότι αυτός είναι ο δρόμος ε, για να βγούμε από τα χρέη. Είναι ψέμα. Στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα το αποτέλεσμα είναι φτώχεια. Δεν δημιουργήθηκε κανένας πλούτος. Και όχι μόνο δεν μειώθηκαν τα χρέη, αλλά αυξήθηκαν κιόλα. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει κανείς να το δει αυτό και να δει ότι αυτή η κατάσταση μόνο βυθίζει περισσότερο στη φτώχεια και στην κρίση αυτές τις χώρες. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που μεταναστεύουν σε άλλες χώρες οι περισσότεροι αναγκάζονται αλλά βεβαίως μπορούν να, να το κάνουν γιατί είναι υποχρεωμένοι, ε, δεν έχουν ανελακτική, αλλά μπορεί να συνεχίσουν να παραμένουν στη χώρα τους και να αγωνίζονται για, για μια ε, κατάσταση για, μια, για την αλλαγή της κατάστασης στην, Ευρωπαϊκή, στην, στη χώρα τους. Εμείς... Ε, τελικά η κατάσταση τι είναι. Οι μετανάστες ε, δημιουργούν πλούτο σε άλλες χώρες και όχι στη δική τους χώρα και αυτό δεν έχει να κάνει με τις δίθεν πολιτικές σύγκλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές που ήρθαν και ευχαριστώ τους ε, ε, συμμετέχοντες. Σας πάμε. Θα τα πούμε σε όλα τα διάφορα σεμινάρια. Directed to your workshop rooms. Okay, so no break. Sorry. <laughs> Not my fault.